Dear I like to start meeting. like to welcome all Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να καλωσορίσω όσους βρίσκονται εδώ και να παρακαλώσω να σταματήσουν οι ομιλίες για να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης, και την έγκριση αυτή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Έχετε την τελική μορφή της σημερινής διάταξης, τη λάβατε την περασμένη Τρίτη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείτε ότι εγκρίνεται. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής διάταξης. Έχω κάποιες ανακοινώσεις να σας ενημερώσω σχετικά με τη συνάντηση της ομάδας εργασίας που ξεχάστηκε εδώ σε αυτή την Επιτροπή γιατί δεν υποβάλλονται συχνά εκθέσει για αυτό το θέμα. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα εργασία για την ερμηνεία και την εφαρμογή τη Διοργανική Συμφωνία για την βελτίωση τη Νομοθεσία. Η τελευταία συνεδρίαση αυτή τη ομάδα εργασία πραγματοποιήθηκε στι 26 Μαρτίου και έγινε μια ανταλλαγή απόψεων για την απλούστευση με τον ε, συνάδελφο από την Κομισιόν, επικεφαλής της μονάδας για την αξιολόγηση, την ε, ρυθμιστική καταλληλότητα και απόδοση, τον κύριο Νόρμπερτ Σάξερ και την κυρία Κάουφμαν που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Γιούρη για την έκθεση Ρίφιτ. Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην ε, Διοργανική Συμφωνία για την Βελτίωση Νομοθεσίας υπήρχαν και αποφάσεις σχετικά με την ε, έναρξη δύο νέων διαπραγματεύσεων. Η μία αφορά την, ε, τα κριτήρια οριοθέτησης για τις κατηγορίες, και τις εκτελεστικές πράξεις. Είχαμε ορίσει δύο εισηγητέ. Ο ένας είναι από τη δική μας επιτροπή, νομίζω είναι ο Ρίτσαρτ Κόμπερτ και ο άλλος είναι ο κύριος Γιώζεφ Σάγερ από την Επιτροπή Γιούρι και ελπίζαμε να ξεκινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις για αυτήν την διοργανική συμφωνία, σύμφωνα και με την ε, διοργανική ε, συμφωνία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστήρηση. Αλλά τίποτα δεν έγινε από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι τον Μάρτιο φέτος. Έτσι λοιπόν, η ΑΦΚΟ και η Γιούρη, οι πρόεδροι δηλαδή των δύο επιτροπών, αποστήλαμε μια επιστολή στον πρόεδρο Ταγιάννη προκειμένου να ασκήσει ποιήση με διπλωματικό τρόπο στους ομολόγους του, στο Συμβούλιο και, και στην Κομισιόν έχει αποσταλεί λοιπόν αυτή η επιστολή και περιμένουμε την απάντηση των άλλων δύο θεσμικών οργάνων. Ελπίζουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει το συντομότερο δυνατό. Έχουμε εμεί ε, βεβαίω οριστικοποιήσει τη δική μα θέση από το 2014 κιόλα. Ελπίζουμε λοιπόν σύντομα να λάβουμε απάντηση από τις, τα άλλα δύο όργανα σχετικά με αυτές τις διαπραγματεύσει. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω όσον αφορά τη διαδικασία του Brexit ότι η διάσκεψη των Προέδρων έχει οριστικοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο αυτό που ε, ονομάστηκε ε, διευθύνουσα ομάδα ε, όπου ε, προετοιμάστηκε το ψήφισμα. το έργο αυτής της ε, ομάδας θα συνεχιστεί και ο, από, το, από το ΕΛΚ εκπροσωπεί, τον, εκπροσωπείται ο κύριος Μπρόκ, ο κύριος Γκουαλτιέρη από τους σοσιαλιστές από τους Πρασίνους είναι ο Φίλιμ Λαμπέτς και η κυρία Τσίμερ από την Γκούε. Ε, συμμετέχει και η Γκούε λοιπόν σε αυτή την ομάδα και ο πρόεδρος της ΑΦΚΟ εκπροσωπεί την επιτροπή μας. Ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε ε, καθήλυνα αρμόδιοι στο τέλος αυτής της διαπραγμάτευσης. Επομένως, συνεχίζει το έργο της αυτό, αυτή η διευθύνουσα επιτροπή να σας ε, ενημερώσω επίσης ότι ο κύριος Μπαρνιέ, όπως μας είχε ε, υποσχεθεί, θα επισκεφτεί την ΑΦΚΟ για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα. Ελπίζω αφού ε, επιτελέσει το έργο της και η ομάδα εργασίας που έχουμε συστήσει. για νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε διάφορες συζητήσεις με τον κύριο Μπαρνιέ. Σε κάθε περίπτωση θα τον προσκαλέσουμε όταν πια συσσωρευτούν τα γεγονότα του επόμενου καιρού για να έχουμε και κάτι να συζητήσουμε. Αυτά και περνάμε με αυτό στο σημείο 3 της σας διάταξης που είναι η έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν δύο συνεισηγητές για αυτήν την έκθεση. Είναι ο Πέντρο Σίλβα Περέρα από τους Σοσιαλιστές και εγώ από το ΕΛΚ να ξεκινήσω εγώ και στη συνέχεια να δώσω το λόγο στον Πέντρο για να κάνουμε την εισήγηση. Έχετε λάβει το έγγραφο εργασίας, εξ όσων γνωρίζω. Να σας υπενθυμίσω όμω κάποια βασικά πράγματα που σχετίζονται με τη διαδικασία ε, γιατί ε, είναι ένα από αυτά τα θέματα όπου η διαδικασία είναι δύσκολη και περίπλοκη για το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η φυτία αυτή, η σύνθεση του Κοινοβουλίου καθορίζεται με βάση την απόφαση του Συμβουλίου του 2013. Σε αυτήν την απόφαση το Συμβούλιο επίσης ζήτησε από το Κοινοβούλιο να υποβάλει πρόταση έως το τέλος του 2016 για ένα σύστημα, μια πρόταση για ένα σύστημα το οποίο στο μέλλον θα ε, επιτρέπει πριν από κάθε ευρωεκλογέ να κατανέμονται οι έδρες μεταξύ των κρατών μελών με δίκαιο, αντικειμενικό ε, και πρακτικά εφαρμόσιμο τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη την ε, αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Αυτό λοιπόν έπρεπε να το είχαμε κάνει ως το τέλος του 2016. Είχαμε ξεκινήσει στην ΑΦΚΟ το σχετικό έργο έγκαιρα. Στη συνέχεια όμως η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως ότου ξεκινήσει η ενεργοποίηση του άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο για ευνόητους λόγους, για κάποιους, για άλλους ίσως λιγότερο ευνόητους. Πάντως αυτή ήταν η απόφαση και στις 6 ε, Απριλίου, μόλις στις 6 Απριλίου, την Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων ξεπάγωσε, αποφάσισε να ξεπαγώσει την διαδικασία και πλέον ε, μπορούμε πια να ε, συνεχίσουμε αυτό το έργο ανοιχτά και όχι ε, και κλεισμένων των θυρών και στους διαδρόμους. Σήμερα λοιπόν θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων για το έγγραφο εργασίας. Δεν είναι έκθεση, ούτε πρόταση έκθεσης ακόμα. Ε, αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα είναι ότι η απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να αναθεωρηθεί πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές του 2019 και θα πρέπει να εγκρίνουμε την ε, συμφωνία αυτή, την απόφαση αυτή ως θεσμικά όργανα αρκετά έγκαιρα ώστε να μπορούν και τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη την απόφαση αυτή κατά την οργάνωση των ευρωεκλογών και φυσικά ε, δεν είναι μόνο τεχνικά δύσκολο θέμα, είναι και πολιτικά ευαίσθητο το θέμα αυτό λόγω των, ε, στο πλαίσιο των εκλογών αλλά και λόγω των πιθανών αλλαγών ε, που επέρχονται από το γεγονός ότι υπάρχει μια πιθανή αποχώρηση κράτους μέλους πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές. Όλα αυτά βεβαίως περιπλέκουν τα πράγματα σαφώς. Η διαδικασία ε, που προτείνουμε ως... είναι η εξή. Εμείς υποβάλλουμε πρόταση ως Κοινοβούλιο, πάει στο Συμβούλιο, εκεί εξετάζεται η πρόταση αυτή ή μπορεί και να μην εξεταστεί και να, ε, το Συμβούλιο να καταλήξει σε μια δική του ε, απόφαση και έπειτα από ομόφωνη απόφαση η απόφαση αυτή του Συμβουλίου στέλνεται στο Ευρωκοινοβούλιο όπου με απλή πλειοψηφία το Κοινοβούλιο δίνει τη συγκατάθεσή του στην απόφαση του Συμβουλίου. Είναι μία από αυτές τις διαδικασίες λοιπόν που απαιτούν έργο από τη δική μας πλευρά, το οποίο πρέπει να υποβάλουμε στο Συμβούλιο, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν και εκείνα να βεβαίως με τη σειρά τους να υποβάλουν σοβαρές τροποποιήσεις ή αλλαγές στη δική μας πρόταση. Εμείς ως Επιτροπή είμαστε αρμόδιοι να υποβάλουμε αυτή την πρόταση αλλά και ο πολιτικά ευαίσθητος χαρακτήρας ε, του θέματος σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και σε πολιτικές ομάδες γιατί η απόφαση για το γιατί θα, μεταξύ άλλων θα πρέπει να αποφασιστεί και το μέγεθος, ο αριθμός των εδρών του Κοινοβουλίου. Οργανώσαμε και μια ακρόαση, κάποιοι θα τη θυμάστε, την, τον Ιανουάριο, με διάφορους εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας περιέγραψαν τα διάφορα μοντέλα που υπάρχουν γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να βρούμε ένα μοντέλο με το οποίο θα μπορέσουμε να ε, αποφύγουμε τις ε, αιματηρές ε, συζητήσεις και διαμάχες πριν από κάθε έτος ευρωεκλογών Εν πάση περιπτώσει, ε, αυτή τη στιγμή αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε είναι να εργαστούμε για αυτό το μοντέλο. Έχουμε λοιπόν αυτό το έγγραφο εργασίας. Θα ακούσουμε τις δικές σας απόψεις σήμερα και στη βάση της συζήτησης που θα γίνει σήμερα θα ετοιμάσουμε την έκθεση. Ε, θα δούμε πόσο, θα χρειαστεί, πόσο χρόνο θα χρειαστούμε γι' αυτό και να υπενθυμίσω επίσης ότι... Ε, η συνθήκη προβλέπει μέγιστο αριθμό εδρών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνθήκη επίσης ε, προβλέπει τα, τα ανώτατα και κατώτατα όρια των εδρών που κατανέμονται ανακράτος μέλος και υπάρχει και η, η συνθήκη επίσης προβλέπει και την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας και ο ορισμός της φθήνουσας αναλογικότητας υπάρχει και στο ψήφισμά μας το 2007 και στο ψήφισμα του Μαρτίου του 2013 όταν και υποβλήθηκε η τελευταία σχετική πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γενικά, λοιπόν, ο ορισμός είναι πολύ γενικόλογος ε, της φθήνουσας αναλογικότητας εννοώ, ε, με πολύ απλούς όρους ε, περιγράφεται η έννοια αυτή. Έχουμε πει ως μπούσουλα στο παρελθόν ότι οι μικρότερες χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες έδρες από ό,τι τους αναλογούν απλά με, μια μαθηματική μέθοδο των τριών. Ε, αυτός όμως είναι, είναι όμως μια πολύ γενική αρχή. Να υπενθυμίσω επίσης ότι το σεμινάριο, το εργαστήριο που είχαμε διοργανώσει, ε, εκεί υπήρξε μια παρουσίαση διαφόρων μοντέλων, τα οποία ε, βεβαίως ε, ωφελούν ή βλάπτουν ε, εντό εισαγωγικών τις, ε, τον αριθμό των εδρών που κατανέμονται σε κάθε χώρα μέλος. Ε, μπορούμε βεβαίως όλα αυτά να τα συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος ε, στο μέλλον, όταν θα είναι καταλληλότερος ο καιρός. Νομίζω ότι σταματήσω εδώ για να δώσω τώρα το λόγο στον Πέδρο, τον συνεισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, υπόθηκαν πολλά. Να ξεκινήσω λέγοντας ε, και εξηγώντα ότι ο σκοπός του εγγράφου εργασίας μας είναι να υπενθυμίσουμε το, τις, τους ισχύοντες νομικούς κανόνες και να υπενθυμίσουμε και τις προηγούμενες συζητήσεις και αποφάσεις που έχουμε λάβει στο θέμα αυτό. Επίσης, θα ήθελα να συνοψίσω κατά κάποιο τρόπο και τις μελέτες και τις συμβολές των εμπειρογνωμών που έχουμε λάβει και να επισημάνω τα βασικά πολιτικά θέματα προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση που θέλουμε να έχουμε σήμερα μαζί σας και στο επόμενο διάστημα. Σκοπός της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνολικά είναι να υποβάλει πρόταση για ένα μόνιμο σύστημα σύμφωνα βεβαίως με τις αρχές, ε, των συνθήκων. Οι συνθήκες ε, καθορίζουν τον ανώτατο αριθμό των εδρών, τα ανώτατα και κατώτατα όρια για κάθε κράτος μέλος και την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας όπως ε, ανέφερθηκε ήδη. Σκοπός μας και καθήκον μας λοιπόν είναι να προσδιορίσουμε τις ε, πιθανές μεθόδους, να συζητήσουμε την πλέον κατάλληλη και να ε, προσδιορίσουμε την πλέον κατάλληλη και θέλω να τονίσω ότι η διαδικασία αυτή προβλεπόταν να ακολουθηθεί πολύ πριν το Brexit. Το Brexit βεβαίως θα επιφέρει κάποιες επιπτώσεις στην διαδικασία που εμείς ε, ε, θα ακολουθήσουμε, αλλά είναι μια συζήτηση την οποία ε, έτσι κι αλλιώ οφείλαμε να κάνουμε σχετικά με τη μόνιμη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τούτων λεχθέντων γνωρίζουμε πλέον ότι Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι οι οποίες είναι συμβατές με την αρχή της ε, ευθύνουσας αναλογικότητας. Κάποιοι λένε ότι είναι 77 στον αριθμό, φαρονικός αριθμός θα έλεγα. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση στο τέλος. Λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις απόψεις των εμπειρογνωμένων, ε, θα πρέπει το σύστημα αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό, αλλά σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ε, ε, λήψη πολιτικής απόφασης. Επίσης, να μην ξεχνούμε ότι η λύση για την, για την κατανομή των εδρών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ισορροπία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για πολλά κράτη-μέλη υπάρχει ένας συμβιβασμός μεταξύ δύο βασικών αρχών στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισότητα μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ισότητα μεταξύ των πολιτών. Φυσικά γνωρίζουμε ότι κάθε αλλαγή στο σύστημα ψηφοφοριών στο Συμβούλιο απαιτεί ε, τροποποίηση συνθήκης. Με βάση αυτό λοιπόν ωστόσο δεν πρέπει να ε, ε, πούμε ότι επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ε, συνθήκη στο άμεσο μέλλον δεν θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αντιστοιχία και η ισοδυναμία των συστημάτων ψηφοφορία στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο θα μα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και δεν θα μα επιτρέψει να έχουμε την καθαρότητα ε, για να λάβουμε τις αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε. Το ε, σύστημα της... Ε, κάποιοι μάλλον θεωρούν ότι το σύστημα της ε, της ενισχυμένης πλειοψηφίας ε, είναι καταστροφικό για, ιδίως για τις μεσαίου μεγέθους χώρους. Γι' αυτό είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, όσον αφορά το σύστημα κατανομής των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία θα τύχει της ομόφωνης υποστήριξης στο Συμβούλιο και η οποία θα είναι αποτέλεσμα πολιτικής συμφωνίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, δεν θα ήταν λογικό να περιμένει κανείς ότι ε, ε, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια ρεαλιστική πολιτική απόφαση. Θα χρειαστεί να συζητηθούν μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι πιθανές επιπτώσεις του Brexit στο μέγεθος του Κοινοβουλίου. Κάποιοι επίσης θέτουν το ζήτημα της ηθαγένειας έναντι του πληθυσμού του εκάστοτε κράτους μέλους όσον αφορά την ε, κατανομή των εδρών και τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Σκοπός του εγγράφου εργασίας λοιπόν είναι να προσδιορίσουμε τα πολιτικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση και νομίζω ότι με το παραδοσιακό μας πνεύμα συνεργασίας θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Αυτό το παραδοσιακό πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ θετικό που το επικαλείστε. Έχουμε πέντε ομιλητές. Ε, Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε όποιος θέλει να πάρει το λόγο στο δηλώσει τώρα. Οκτώ ομιλητές πλέον στη λίστα. Για 35 Πέντε περίπου λεπτά, Τέσσερα λεπτά κατά άτομο. Και Βίλαντ πρώτος. Φρέντα. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι θα ήμουν πρώτος. Ε, δεν ήθελα να πάρω τη θέση κανένα. Λοιπόν, στο έγγραφο εργασίας ε, διατυπώνονται διάφορα ερωτήματα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει άλλο ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Στο έγγραφο ε, περιγράφεται ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και η διαδικασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο όρος δημοκρατικό έλλειμμα είναι ένας όρος που τον έχουμε ακούσει πάρα πολύ και ε, περιόδους ε, που το Κοινοβούλιο ακόμα δεν είχε ακόμα αρμοδιότητες. Νομίζω όμως ότι δημοκρατικό έλλειμμα μπορεί να δημιουργηθεί ε, και σε περίπτωση που ε, το 75% των ψηφοφόρων δεν αντιστοιχούν στο 75% των εκπροσώπων των πολιτών. Επίσης, θέλω να πω ως Γερμανός ότι χρειαζόμαστε μία φόρμουλα ώστε να μπορούμε να πούμε ε, και στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας μου ότι οι έδρες δεν κατανόμονται με αυθαίρετο τρόπο. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σχετική προβλεψιμότητα για το σύστημα αυτό. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο, θεωρώντας δεδομένο το Brexit βεβαίως, σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα έχει πολύ λιγότερα χρήματα στη διάθεσή του. Το να περιμένει λοιπόν κανείς ότι αυτές οι έδρες που θα μείνουν κενές θα κατανεμηθούν στους άλλους, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι τέτοιο δεδομένο Νομίζω ότι ο σωστός τρόπος εργασίας είναι να πούμε ότι οι Βρετανοί εξακολουθούν να είναι μέλη και η σύνθεση του επόμενου κοινοβουλίου θα υπολογιστεί σαν να παραμένει κανονικά η Βρετανία χώρα μέλος της Ένωσης. Και αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε αυτές οι θέσεις του μάλλον θα ε, μείνουν κενές, αδιάθετες. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ε, εξοικονομήσουμε και χρήματα, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα φανεί σαν να μοιράζουμε τη λία μεταξύ μας. Αυτά είναι τα δύο πρώτα θέματα που ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, όσον αφορά τη φτύνουσα αναλογικότητα, πρέπει να πούμε το εξής. Όποιο και είναι το σύστημα κατανομής, μαθηματικά, η τελευταία έδρα που κατανέμεται πάντοτε μπορεί να ε, δημιουργήσει αδικία. Αν έχετε 8 χώρες με 3 εκατομμύρια κατοίκους, όλοι έχουν ε, περίπου τις ίδιες, τα, ίδια υπόλοιπα και θα πρέπει να, να κατανεμηθεί και τότε σε αυτή την περίπτωση η μικρότερη χώρα δεν θα πάρει έδρα και έτσι δημιουργείται μια δυσαναλογία. Αν το σκεφτείτε, μια αδικία δηλαδή του εκλογικού συστήματος. Δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει αυτός. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ε, ε, ε υπάρξει ένα αμάλγαμα και της απλής και της ενισχυμένης πλειοψηφίας. Νομίζω ότι θεωρητικά μετά την ε, κατανομή των εδρών μπορεί κάποια, κάποια χώρα να έχει και μηδέν έδρες αρχικά στην πρώτη κατανομή και στη συνέχεια να μπορεί μια χώρα ε, να με βάση τον τύπο που προβλέπετε να ε, κατανέμονται σε κάθε χώρα 6 έως 90 έδρες και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα να καταλήγουν σε μια αναλογική κατανομή. Αυτό βεβαίως ε, θα δημιουργήσει ε, σοβαρές αλλαγές. αλλαγές φυσικά δεν μπορεί να ε, παραμείνει η κατάσταση με τη Γαλλία όπως έχει αυτή τη στιγμή. Είναι παραβίαση της αρχής της θύνωσης αναλογικότητας αυτό που συμβαίνει με τη Γαλλία. Επίσης δεν μπορούμε χώρες που έχουν 20 έδρες να τους πάρουμε το 10% των εδρών τους πίσω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει στην νέα ε, φόρμουλα και τη νέα μέθοδο υπολογισμού που θα καθοριστεί και μια μέθοδος, μέθοδος απορρόφησης των κραδασμών αυτών. Δέκα εκατομμύρια. Οι χώρες που έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους δεν θα πρέπει να χάσουν περισσότερο από μία έδρα ό,τι και να γίνει. Γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να, να εξασφαλίσουμε μια σταδιακή εισαγωγή σε ένα νέο σύστημα το οποίο θα τελειοποιείται κιόλα με την πάροδο του χρόνου, αλλά θα υπάρχει αυτό που είπα στην αρχή, προβλεψιμότητα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για έναν, επίσης, ε, για έναν ακόμη λόγο. Ο τύπος πρέπει να ε, εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν παραβιάσεις. Γιατί αν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα δεν θα βρεθούμε ποτέ ξανά στην ε, δυσάρεστη θέση που βρεθήκαμε την τελευταία φορά να ψηφίσουμε ε, μεταξύ δύο χωρών και να καταψηφίσουμε δηλαδή μία χώρα. Αν ε, υπήρχε σαφής μαθηματικός τύπος τότε δεν ε, υπάρχει περίπτωση και εμείς να βρεθούμε σε αυτή τη μέγενη του να καλούμαστε πολιτικά στην ουσία να αποφασίσουμε ποιος θα ωφεληθεί και ποιος όχι. Η κυρία Jones, όχι η κυρία Τζέιμς. Thank you very much, Madam Chair. Τέσσερις παρατηρήσεις έχω να κάνω και θα ήθελα και απαντήσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το μέγεθος του πληθυσμού, πάρτε, ε, βγάλτε το Ηνωμένο Βασίλειο από την εικόνα για τους γνωστούς λόγους. Ε, εμείς έχουμε απογραφεί κάθε 10 χρόνια. Η Γαλλία, από την άλλη μεριά, έχει ε, μια ε, ετήσια απογραφή βασισμένη σε δείγμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα φτάσουμε σε μια κοινή εικόνα του ποιος είναι ο πληθυσμός σε κάθε χώρα. Δεύτερη παρατήρηση. Το πού βρίσκονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής και το πώς είναι δυνατόν να μην μετρούνται δύο φορές. Ε, το θέμα της μετανάστευσης ήταν επίμαχο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν 900.000 Πολωνοί υπηκόοι που ε, ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πού όμως ψηφίζουν. Ψηφίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο, στην Πολωνία και πού θα καταμετρηθούν σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών. Τρίτη παρατήρηση. Ε, πώληση διαβατηρίων ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξέρουμε ότι ε, υπάρχει αυτό το φαινόμενο και θέλω να δω τι δικαιώματα δίνει σε αυτούς που αγοράζουν διαβατήριο. Ε, και τέταρτον, ο κ. Φερχόφστατ έχει ένα παράξενο όραμα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή υπηκότητα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Και το αντίστροφο όμως μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να αποκτήσουν την υπηκότητα του Ηνωμένου Βασιλείου ή μια άλλη. Πώς αυτό θα ληφθεί υπόψη μέσα στα μοντέλα τα οποία συζητούμε. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να κάνω μια σκέψη ό,τι αφορά την αρχή. Η κατανομή των εδρών. Θα πρέπει να γίνει μέσα σε συνθήκες λίγο ιδιαίτερες. Αυτή τη στιγμή υφίσταται ένα δημοκρατικό έλλειμμα και μια έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών μας ε, σε σχέση με τα θεσμικά όργανα και τους πολιτικούς. Η απόφαση λοιπόν κατανομής θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τα ερωτηματικά που έχουν οι πολίτες μας στο μυαλό τους. Θα πρέπει δηλαδή η πρότασή μας να είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες των πολιτών μας. Τώρα, η διαδικασία αυτή δεν είναι καινούρια. Το 2013-2014 ήδη κάναμε μια προσπάθεια να βρούμε μια μόνιμη σε εισαγωγικά λύση. Τώρα με το Brexit αυτή η μόνιμη χτεσινή λύση δεν μας κάνει για αύριο. Όλα τα θεωρητικά, μαθηματικά μοντέλα τα οποία συζητήσαμε στην περασμένη θητεία μας, αλλά και τον Ιανουάριο στο σεμινάριό μας, είναι δυσνόητα. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς πώς λειτουργούν και δεν μπορούν να μας χρησιμεύσουν για να τα παρουσιάσουμε στην κοινή γνώμη. δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στους πολίτες και να εξηγήσουμε και τη λογική τους. Ε, εμείς ε, καταφύγαμε πριν από μερικά χρόνια στο συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας στην Καλσρούη και μας είπαν οι συνταγματικοί δικαστές ότι περιμένουν από τους κανόνες του Κοινοβουλίου μία σαφή και αντιπροσωπευτική εικόνα της κατανομής του πληθυσμού όταν κατανομούμε τις έδρες. Και βέβαια αυτό έχει σχέση και με την κατανομή των ψήφων, ε, δηλαδή το θέμα των πολιτικών κομμάτων, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και πώς συνδέονται με τα εθνικά πολιτικά κόμματα. Καταλαβαίνετε, ε, το θέμα είναι πολύ περίπλοκο εννοώ ε, και δεν είναι περίπλοκο όχι μόνο τεχνικά αλλά και ως ε, και ως αρχές οι οποίες θα πρέπει να το διέπουν. Ακόμα και η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας είναι δύσκολο να περιγραφεί. Τώρα, ας είμαστε μετριοπαθείς. Γιατί ας μην θεωρήσουμε ότι είναι δεδομένο το Brexit αυτή τη στιγμή. Ας ε, μην θεωρήσουμε ότι οι έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ελεύθερες τη στιγμή που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε ε, ή στις επόμενες εκλογές μπορεί να έχουμε και καινούρια μέλη Οπότε ενδεχομένως δεν θα έπρεπε ε, ήδη να καλύψουμε και τις 751 έδρες του Κοινοβουλίου, έχοντας στο μυαλό μας, λέω, ότι μπορεί να ενταχθεί και κάποιο άλλο κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει Καταρχήν να αποφασίσουμε αν θα εφαρμόσουμε το κριτήριο DON'T ή κάποιο άλλο για την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο. Αλλά οποιοδήποτε τρόπο και αν διαλέξουμε, οποιοδήποτε μέθοδο και να διαλέξουμε, θα πρέπει να μπορούμε να την εξηγήσουμε στους πολίτες μας. Υπάρχουν διπλές πλειοψηφίες, διπλές πλειοψηφίες υπάρχουν ε, εθνικές ιδιαιτερότητες, οτιδήποτε λάβουμε υπόψη μας θα πρέπει να μπορούμε να το εξηγήσουμε. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά πρέπει να είμαστε πιο ε, γενναίοι, πιο τολμηροί στις αποφάσεις μας. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όχι αυτό το οποίο εύκολα θα δεχτεί το Συμβούλιο, να μην αυτολογοκριθούμε, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μιλήσει για παράδειγμα για ευρωπαϊκές λίστες στις εκλογές. Ε, μήπως πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε περισσότερο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από την Ευρώπη των 27. Να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο για το ε, απότερο μέλλον. Τελικά η εξουσία βρίσκεται στα χέρια των πολιτών μας. Ο κυρίαρχος είναι ο λαός. Και αυτό θα αποφασίσει. Um, Θέλω να κάνω κάποιες, ε, κάποια πολιτικά σχόλια, κάποιες πολιτικές παρατηρήσεις. Ε, κάποιοι από εσά γνωρίζετε ότι είμαι βετεράνος εδώ και θυμάμαι και τις παλιότερες συζητήσεις και αυτό που θυμάμαι είναι ότι το κάθε μαθηματικό μοντέλο, όσο τέλειο ή ατελές και να είναι, έχει κάποιες πολιτικές υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται. Δηλαδή, στη βάση κάθε μοντέλου είναι μια πολιτική απόφαση η οποία εξειδικεύεται μέσω μιας μαθηματικής φόρμουλας. Οπότε κάθε μαθηματικό μοντέλο έχει κάποιες επιδράσεις, τις οποίες εμείς εκ των προτέρων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μ' αρέσει ο συμβασμός της προηγούμενης θητείας, του, ο, ο συμβασμός Τσαρκόφσκι που λέγαμε, ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα έπρεπε να χάσει περισσότερο από μία ε, έδρα Αναγνωρίζω το πρόβλημα τη Γαλλία βέβαια, το οποίο αναφέρατε πολύ. Σω εκεί χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη λύση. Άλλε παρατηρήσει που έχουν να κάνουν είναι εξή. Πληθυσμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει τους πολίτες και πρέπει να γνωρίζουμε ποιο ποσοστό του πληθυσμού είναι υπήκοοι ε, τρίτων χωρών. Γιατί αυτό θα αλλοιώσει, θα αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί η αύξηση του πληθυσμού σε κάποια κράτη-μέλη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε πολίτες τρίτων χωρών. Έτσι. Αν τους λάβουμε όλους υπόψη ενός πληθυσμού της χώρας, τότε δεν εκπροσωπεί το κοινοβούλιο μόνο των ευρωπαϊκού, τους ευρωπαϊκούς λαούς. Και το αντίστροφο. Δεν έχω σαφή στοιχεία αλλά περίπου 20-25 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν σε χώρα που δεν είναι δική τους. Πώς εκπροσωπούνται αυτοί, από ποιον. Από ποιον πρέπει να εκπροσωπούνται. Σε παλιότερες συζητήσεις εδώ πέρα είχα πει ότι εγώ προσωπικά δύσκολα μπορώ να φανταστώ πως ο Νάιτζελ Φάρατζ μπορεί να αντιπροσωπεύει τους Πολωνούς που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν ο πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, το τον οποίο θα λάβουμε εμεί υπόψη για την κατανομή των εδρών, θα περιλαμβάνει όχι του Πολωνού αυτού. Και το ίδιο ισχύει και για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτοί οι πολίτε που ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν σε χώρα που δεν είναι δική του, από ποιον εκπροσωπούνται. Άρα, μήπω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη του υπηκόου και όχι τον πληθυσμό. Αυτό βέβαια έχει άλλα αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Το τελευταίο μου παρατήρηση. Η μετανάστευση είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Είναι ε, νούμερα τα οποία συνεχώ αλλάζουν, ρευστά νούμερα. Μετακινήσει πληθυσμό λαμβάνουν χώρα διαρκώς. Οποιοδήποτε σύστημα και αν ε, επιλέξουμε θα πρέπει να είναι δυναμικό. Δεν θα ήθελα ενδεχομένως να καθορίσουμε με σταθερό τρόπο τις ε, έδρες και μετά από 4, 5, 10 χρόνια να ξανασυζητάμε ποιο πρέπει να είναι το μόνιμο σύστημα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ένα μόνιμο σύστημα είναι η λύση στο πρόβλημά μας. Αυτό βέβαια το βλέπω εγώ, ίσως δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει κανείς σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Πάλο Ράνσελ. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχάς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο και στο σύστημα κατανομής των εδρών ε, στο Κοινοβούλιο. Και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στον κύριο Φωσκούλα όταν ακριβώς ε, κλήθηνε να μιλήσω για αυτό το θέμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης. Διότι είναι πολύ σαφές ότι αν στο Συμβούλιο έχουμε ομοσπονδιακό σύστημα όπου κάθε κράτος έχει μία ψήφο, εδώ μπορούμε να έχουμε αναλογικό σύστημα με διόρθωση μόνο για τα πολύ πολύ μικρά κράτη. Ωστόσο, επειδή στο Συμβούλιο έχουμε ένα σύστημα ψήφων όπου ο πληθυσμός βαραίνει, τότε φυσιολογικά εδώ θα, πρέπει, θα έχει σημασία η ιδιότητα πολίτη ή όχι. Το συνταγματικό δικαστήριο Τη Γερμανία δεν είναι δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουμε κάτι που αποφασίζει εκείνο. Όμω αν έχουμε σύστημα ομοσπονδιακού τύπου όπω η Γερμανία που δίνει τρεις έδρε στην Άνω Βουλή και έξι στις μεγάλες τότε μπορούμε να, να αφήσουμε μια τέτοια αναλογία και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν θέλουμε να μιμηθούμε αυτό το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε μπορούμε να έχουμε ένα αναλογικό σύστημα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά την εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και αλλαγή της συνθήκης και αλλαγές στο Συμβούλιο. Όλες οι αλλαγές λοιπόν θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά. Αυτό είναι το πρώτο μου επιχείρημα. Το δεύτερο είναι το εξής. Πιστεύω ότι με το Brexit έχουμε μια ευκαιρία να ολοκληρώσουμε και τα κριτήρια χωρίς να δημιουργήσουμε πολιτικό πρόβλημα στα κράτη που θα πρέπει να χάσουν πολλές έδρες αν θέλαμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Η σύστασή μου θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε μόνο 23 βουλευτές, ευρωβουλευτές και αυτό πιστεύω πως θα αρκεί για να γίνει η ανακατανομή εδρών που θα σέβεται την ανταλογικότητα ΔΕΓΡΕΦ και δεν θα δημιουργεί την ευθύνουσα αναλογικότητα και θα είναι όλα, όλοι ευχαριστημένοι. Έχουμε δύο, δύο λοιπόν επίπεδα. Από τη μια έχουμε πολιτική διαπραγμάτευση που θα είναι πολύ εύκολο να δώσουμε στην Γαλλία, στην Ισπανία, πιθανότατα ε, στι κατοχώρε, στην Ιρλανδία, κάποιε ε, έδρε ώστε να υπάρχει δίκαιη φθήνουσα αναλογικότητα, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι πολιτική αναδιαπραγμάτευση και όχι ένα μόνιμο σύστημα, αλλά ένα μόνιμο σύστημα είναι επίσης πολυ, πολιτικού χαρακτήρα, γιατί δεν υπάρχει ε, ουδέτερη μαθηματική ουδέτερο μαθηματικό τύπο. Το έχουμε αυτό συζητήσει πολύ έντονα και στην προηγούμενη θητεία. Και άλλη μια δυνατότητα είναι να εξετάσουμε έναν από αυτού του τύπου, ιδιαίτερα το τελευταίο που περιλαμβάνει δύο κριτήρια νομίζω ότι είναι ίσως μια λύση εάν δηλαδή χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους 23 ευρωβουλευτές 21 εντάξει αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε Πάντως, είτε πολιτική διαπραγμάτευση, είτε ένας μόνιμος τύπος, τώρα με το Brexit έχουμε την ευκαιρία επιτέλους να ε, θέσουμε σε εφαρμογή την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, νομίζω. Επίσης θα θέλω να δηλώσω πως είμαι πολύ σε μεγάλο βαθμό βέβαιος ότι τα κράτη μεσαίου μεγέθους, δηλαδή ανάμεσα στη Λουθιανία και τη Ρουμανία δεν θα δεχτούν σύστημα όπου απλώς θα συνθλιβούν γιατί οι προτάσεις που προέρχονται από μεγαλύτερα κράτη-μέλη συνήθως ε, συμφωνούν με αυτή την ιδέα του να σεβαστούν τα μικρά κράτη αλλά προσπαθούν να συνθλίψουν τα μεσαία κράτη. Αυτό σας το λέω γιατί όπως και την τελευταία φορά έχουμε άτυπες επαφές με τα κράτη-μέλη και έχουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό ε, ευρωπαϊκού πληθυσμού και αυτό θα είναι κόκκινη γραμμή. Γι' αυτό είμαι πολύ βέβαιος. Ευχαριστώ, κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές για το έγγραφο εργασίας που νομίζω ότι θέτει τα σωστά ερωτήματα. Ε, Θεωρώ ότι η, πρόεδρο πρόεδρος έχει μεν δίκιο λέγοντας ότι το έργο ε, από πλευράς Κοινοβουλίου είχε ξεκινήσει πολύ πριν το Brexit και το σχετικό δημοψήφισμα. Από την άλλη πλευρά όμως η ευρωπαϊκή ε, κοινή γνώμη θα έχει αυτό και μόνο στο επίκεντρό της. Γιατί σε κάθε χώρα τα βλέμματα θα στραφούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πώς θα χειριστούμε αυτή την υπόθεση. Θα καταφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μειώσει τους ε, βουλευτές του ή θα κατανείμει τις ε, έδρες των Βρετανών στις άλλες χώρες. Νομίζω ότι ε, θα είναι το κυρίαρχο θέμα στην ενόψη των επόμενων ευρωεκλογών. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε πολιτικά, να αποφύγουμε ε, λάθη και να αποφύγουμε να οριστικοποιήσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι μόνιμο και ενδεχομένως θα ε, κατανείμει ακόμη και τις ε, Βρετανικές έδρες στις άλλες χώρες. Πρώτον, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κανείς δεν ξέρει σε δύο χρόνια πώς θα έχει διαμορφωθεί η πολιτική κατάσταση και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το έργο μας με διάφορες δυνητικές πιθανές εκδοχές. Ε, θα υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο με 751, ένα σχέδιο όπως το περιέγραψε ο συνάδελφος Ρανζέλ, ε, με λιγότερους, με 723, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο θα λέει ότι εντάξει, αποχωρούν οι Βρετανοί, κάτι που μας επιτρέπει να εξοικονομήσουμε ε, έδρες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μειωθεί δηλαδή η σύνθεση, ο αριθμός των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά 73. Θα πρέπει και τα τρία εναλλακτικά σχέδια να μείνουν ανοιχτά και να ληφθούν υπόψη και στην πολιτική διαπραγμάτευση που θα γίνει από εδώ και στο εξή. Γιατί νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να οριστικοποιήσουμε από τώρα, εν ώψη των ευρωεκλογών, ε, την, ε, τον οριστικό αριθμό, εν πάση περιπτώσει, των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, θα πρέπει να μην ανοιχτά τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια και να μην αρχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας ε, όπως είπα, εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί κάτι τέτοιο θα κυριαρχήσει, στην, ε, θα κυριαρχήσει στη συζήτηση που θα γίνει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σοντόφσκι. Νομίζω ότι αφετηρία μας θα πρέπει να είναι ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι έδρες της Βρετανίας. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει 73 έδρες λιγότερες. Κάτι τέτοιο θα είναι διαφανές, θα είναι απόλυτα κατανοητό από τους πολίτες, και θα αποστείλει και ένα μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να δρά με πιο οικονομικό τρόπο από ό,τι το έκανε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι οι συνεισηγητές θα πρέπει να υποβάλουν μια καινοτόμα πρόταση για την κατανομή των εδρών και η λύση αυτή βεβαίως θα πρέπει να εκπληρώνει και τις αρχές της συνθήκης και να συνδυάζεται και με τον τροποποιημένο τρόπο ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Ως αφετηρία λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να μην κατανεμηθούν οι έδρες των Βρετανών στα άλλα κράτη-μέλη, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη στεναρή υποστήριξη σε μια τέτοια ε, επιλογή. Νομίζω ότι οι συνεισηγητές οφείλουν να υποβάλουν επιχειρησιακού χαρακτήρα ε, προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να τεθούν σε συζήτηση. Κύριος Κόμμεντ, ευχαριστώ. Το πρώτο που θέλω να θέσω είναι το ζήτημα του timing, του χρονισμού. Γιατί όποια και αν είναι η πρότασή μας θα πρέπει να τύχει ε, ομόφωνης ε, από το Συμβούλιο και στη συνέχεια να επιστρέψει σε εμά και ταυτόχρονα να δοθεί και ο απαραίτητο χρόνος στα εθνικά κοινοβούλια ώστε να καθορίσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες ή άλλα σχετικά θέματα που μπορούν να ε, ε, σχετίζονται με το θέμα. Έχουμε ήδη χάσει πάρα πολύ χρόνο. Ό,τι και αν είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι το Brexit θα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και τουλάχιστον μια υποσημείωση η οποία θα λέει ότι σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση ή αλλαγή γνώμης από το Ηνωμένο θα πρέπει και αυτοί, αυτές οι πιθανότητες να καλύπτονται από τη δική μας πρόταση. Βασιζόμενοι λοιπόν όμως και υποθέτοντας ότι ε, το Brexit θα ολοκληρωθεί και δεν είναι φυσικά δική μου δουλειά να ε, αποφασίσω θα έλεγα βάσει της πείρας μου ότι δεν είναι απαραίτητο να αναδιανεμηθούν όλες οι έδρες προκειμένου να καλύπτονται μεταξύ των κρατών μελών το ανώτατο όριο των ε, εδρών. Ιστορικά λέγαμε ότι 700, είναι η, ο μέγιστος αριθμός ε, των ευρωβουλευτών. Κάτι τέτοιο μάλιστα είχαμε προτείνει εμείς οι ίδιοι ε, πριν από 15-20 χρόνια. Τα κράτη-μέλη ήταν εκείνα που προσθέτοντας από εδώ και από εκεί διάφορα ε, μέλη ε, καταλήξαμε να ε, είμαστε 751. Τα κτίρια μας χτίστηκαν με βάση ε, την υπόθεση ότι οι ευρωβουλευτές θα ήταν 700. Γι' αυτό και έχουμε διάφορα προβλήματα τώρα πια. Πρόταση μου θα ήταν λοιπόν να μην αναδιανεμηθούν οι θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή να αναδιανεμηθούν μόνο εκείνες ε, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώνεται καλύτερα η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Ε, κάτι τέτοιο βεβαίως πάλι θα μας φέρει στους 700 ευρωβουλευτές όπως και είχαμε πολύ αρχικά προβλέψει. Για το 2024 ωστόσο, που θα ξανά έχουμε ευρωεκλογέ, μπορεί να ε, προβλέψει κανείς ότι μπορεί να είμαστε και περισσότεροι, περισσότερα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει προσχωρήσει το, ευρω, ε, το Μαυροβούνιο, ε, που θα πάρει βέβαια έξι έδρες, όχι παραπάνω, αλλά και πάλι θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του και αυτήν την πιθανότητα. Τώρα, Ω προ τη σύνδεση με το σύστημα ψηφοφορία του Συμβουλίου. Σε ε, παραδοσιακά συστήματα με δύο βουλές υπάρχει ε, η, ισότητα μεταξύ των μελών, των κρατών μελών μιας ομοσπονδίας και υπάρχει και η αρχή της ισότητας των πολιτών. Στο δικό μας σύστημα υπάρχει ε, ένα ε, διπλό σύστημα ψηφοφορίας. Ένα που σχετίζεται με, τη, με, τον πληθυσμό της κάθε χώρας και ένα που σχετίζεται και πηγάζει από την αρχή της ισότητας με των κρατών μελών. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αλλάξει γιατί απαιτεί αλλαγή τροποποίηση της συνθήκης. Αυτό είναι δεδομένο και γι' αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αυτήν την φθήνουσα αναλογικότητα. Είναι με ένα αναλογική δηλαδή η κατανομή των εδρών, αλλά με, ένα μεγαλύτερο βάρος ε, προς όφελος των μικρότερων χωρών. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει διασύνδεση με το σύστημα ψηφοφορίας του Συμβουλίου. Εκτός αν ε, επιχειρηματολογεί κανείς ότι στο Συμβούλιο οι μεσαίες χώρες είναι αυτές που χάνουν. Γιατί δεν έχουν αρκετά μεγάλο πληθυσμό ώστε να βαραίνει ε, ο πληθυσμός τους στην, ε, στις ψήφους τους και ταυτόχρονα ε, έχουν και τον ίδιο αριθμό ψήφων ως, όπως και τα μικρά. Δηλαδή τα, τα μικρά κράτη-μέλη ωφελούνται γιατί έχουν και αυτά μία ψήφο, τα μεγάλα κράτη-μέλη ωφελούνται λόγω του μεγάλου πληθυσμού τους, πληθυσμού τους, τα μεσαία είναι αυτά που αδικούνται. Καταλαών, κατανοώ αυτό το επιχείρημα μεν, αλλά υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία που να ε, στηρίζουν ένα τέτοιο επιχείρημα και αν ναι, από εκεί και πέρα βεβαίως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε εδώ. Αλλά νομίζω ότι ε, το καλύτερο θα ήταν εδώ να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις λιγότερες ε, παραβολικές ε, φόρμουλες προκειμένου να κατανέμονται οι έδρες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ναι, ότι πρέπει να γίνουν οι προσαρμογές χωρίς να λάβουμε υπόψη τις έδρες των Βρετανών. Και όχι γιατί είναι δυνατόν να μπλοκάρουμε το Brexit, όχι, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αυταπάτη, αλλά απλά και μόνο επειδή το ανώτατο όριο των 751 εδρών αναφέρεται στη συνθήκη. Άρα πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον μια ελπίδα σε άλλους ότι θα μπορέσουν να μπουν στην Ένωση χωρίς να, να χρειάζεται αλλαγή συνθήκων. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια κάπως απεσιόδοξη εικόνα στα πέντε σενάρια που παρουσίασε ο αγαπητός Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Μιλάμε για 2025 για μια Ένωση των 27. Πράγμα που σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα υπάρξει νέο μέλος. Ακόμα ούτε καν το Μαυροβούνιο. Ξέρω ότι αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη και σχεδόν ομόφωνη ότι δεν ε, πρέπει να γίνει άλλη διεύρυνση. Εγώ είμαι εξ αυτών που πιστεύουν τη δυνατότητα και τη σημασία των διευρύνσεων πριν το 2025. Ε, Επίση, δεν πιστεύω πως πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε περισσότερο το Συμβούλιο. Χοντρικά μπορεί να βλέπουμε ε, στο Συμβούλιο μια ανοβουλή, δεύτερο σώμα, αλλά δεν θα πρέπει να, βρούμε, να, να στραφούμε προς αυτό που υπάρχει σε κάποια κράτη, δηλαδή το σύστημα των συμμετρικών δύο βουλών. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η συμμετρία ε, στο Συμβούλιο αν το θεωρήσουμε ως ένα άλλο σώμα. Θα πρέπει γι' αυτό να επικρατεί διαφορετική λογική εδώ στο Κοινοβούλιο από αυτή που επικρατεί στο Συμβούλιο. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Είμαι υπέρ της διατήρησης μιας τέτοιας διαφοράς ασυμμετρίας και όχι υπέρ της ιδέας του να υπάρξει περαιτέρω προσέγγιση. Τώρα, όσον αφορά αυτή την υπόθεση που αφορά τους κατοίκους που διαμένουν ή τους ε, υπηκόους. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει να υπολογίσουμε με τον πληθυσμό, που, με τους κατοίκους βασικά, γιατί δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε τη δυνατότητα του κάθε Ευρωπαίου, πέρα από το που είναι η κατοικία του, η δηλωμένη κατοικία του, κάποιες εβδομάδες πριν, ανάμεσα να μπορέσει να διαλέξει ανάμεσα στη χώρα προέλευσής του και τη χώρα κατοικία του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τελευταία στιγμή τέτοιες προσαρμογές όσον αφορά την εκλογική μάζα σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την επιλογή που πρέπει να έχουν και να διατηρήσουν οι πολίτες. Δεν μπορούμε να αυτόν, την ελευθερία ε, να, αυτή να την περιορίσουμε. Ο κάθε μας πολίτης μπορεί να ψηφίσει είτε εκεί όπου διαμένει, είτε στη χώρα προέλευσής του. Και τέλος, συμφωνώ με τη συνάδελφο που μιλούσε για αυτή την παράξενη ιδέα του κύριου Φερχάφστατ να εφεύρουμε δηλαδή και μια ημι, ημι δυνατότητα πολίτη, κάτι μεσοβέζικο, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχω καταλάβει και μάλιστα με ανησυχεί ακόμη περισσότερο, γιατί, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Φερχόφστατ μιλάει στο όνομα του Κοινοβουλίου χωρίς να έχει όμως από ό,τι ξέρω κάποια εντολή για να λέει τέτοια πράγματα. Είναι κάτι το χαοτικό και το ανεξήγητο. Δεν μπορούμε να το... Είναι μια ελεύθερη δημαγωγία, πολύ μυστήρια και πολύ ανησυχητική. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Μάιτε έχει το λόγο. Ε, λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω σε όσους μίλησαν για τον κύριο Φερχόφστερ και τον ανέφεραν. Δεν είμαι και ειδική. Ζήτησα το λόγο. Α, να επαναλάβω. Συγγνώμη. Για όσου μίλησαν για τον πρόεδρο της ομάδα μου που δεν είναι παρόν, ε, ε, ήθελα να σας πω ότι δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματός του. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα πάρετε μια απάντηση, ή θα μπορέσετε να τα σχολιάσετε ε, ε, μπροστά του ε, και ζωντανά. Απ' την άλλη μεριά δεν είμαι και ειδική σε θέματα εκλογικά και δεν ήμουνα καν ευρωβουλευτής το 2013. Όμως, έχω να πω τα εξής. Η κυρία Σιλβί Γκυλιάρ μου είπε να σας εκφράσω το ενδιαφέρον της για το θέμα αυτό και να μιλήσω για το θέμα των ευρωπαϊκών ληστών. Μιλήσατε για πάρα πολλά άλλα θέματα, αλλά η κυρία Γκυγιάρ θέλει να σας υπογραμμίσω το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Λίστας το οποίο θέλει να αναπτύξει και να αναπτύξουμε στο μέλλον. συζήτηση τα σχόλια σας κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ ποιοτικά, η συζήτηση πολύ καλή. Ωραία, αν υπάρχουν ομιλητές να δώσω το λόγο στον Πέντρο. Κύριος Περέιρα. Έχω τα εξή σχόλια. Συμφωνώ με εκείνους που ανέφεραν πως χρειαζόμαστε ένα δίκαιο, μια δίκαιη αντικειμενική και ε, κατανοητή κατανομή και λύση. Η αρχική ιδέα ήταν να έχουμε ένα μαθηματικό τύπο, ένα μόνιμο σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί ανεξαρτήτως του αριθμού των κρατών μελών. Οπότε δεν είναι καλό το επιχείρημα να μην κατανείμουμε, να μην διανύμουμε τις ελεύθερες έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να τις κρατήσουμε για κάποιο μελλοντικό κράτος μέρος. Όχι. Ο, η ίδια φόρμουλα που θα επιλέξουμε θα χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον ακόμα και όταν έχουμε καινούργια κράτη-μέλη. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλλειμμα στο οποίο αναφέρθηκαν κάποιοι. Το, επιχείρημα, το πολιτικό αυτό επιχείρημα είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνέπειες των αλλαγών που βλέπουμε στη συζήτηση περί αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας στα θεσμικά όργανα. Βλέπουμε ε, σημαντικές αλλαγές στο status quo. Κάποιες χώρες θα αν κάποιες χώρες ε, δουν ότι η αντιπροσώπευσή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μειώνεται δραματικά, αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ως αύξηση του δημοκρατικού ελλείμματος. Τέλος, ό,τι αφορά το μέγεθος του Κοινοβουλίου και τη σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα ψηφοφοριών του Συμβουλίου και στην κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω το εξή για αυτό το ζήτημα. Ας αντιληφθούμε αυτή τη σύνδεση, διότι εξηγεί και το επίπεδο αντίστασης, το βαθμό αντίστασης ε, σε ό,τι αφορά την πλήρη εφαρμογή της αρχής της φθήνουσας αναλογικότητας. Γιατί η λύση που έχουμε χρησιμοποιήσει, γιατί χρειάζεται μια ρεαλιστική ε, λύση, γιατί πολλά κράτη-μέλη βλέπουν ότι βλέπουν, ε, θεωρούν προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζεται η ψήφος τους στο Συμβούλιο σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζεται η αντιπροσωπευτικότητά τους στο Κοινοβούλιο. Όμως, αλλαγή του αριθμού των μελών θα απαιτούσε αλλαγή συνθήκες. Ε, αυτό το έχει πει το Συμβούλιο, έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά, Ας καταλάβουμε γιατί δεν είναι πολιτικός δυνατή μια σημαντική αλλαγή στο σημερινό status quo. Γιατί πολλά κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη θα είχαν ε, πάρα πολύ ισχυρές αντιδράσεις. Οπότε χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική, λειτουργική λύση από πολιτικής πλευράς. Θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Κατά την άποψή μου, ένα τμήμα τουλάχιστον των εδρών του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ανακατανεμηθεί. Αυτό είναι σημαντικό για να βρούμε μια πολιτική λύση στο πρόβλημα. Γιατί αλλιώς μπορούμε να συζητάμε μαθηματικούς τύπους, να συζητάμε για τις επιθυμίες μας, τις ευχές μας, αλλά στην πράξη θα είναι πολύ δύσκολο χωρίς αυτές τις έδρες να καταλήξουμε σε πολιτική συνένεση. Ευχαριστώ. Προς τους συναδέλφους όπως η Μάιτε και άλλοι που ε, έχουν στο μυαλό τους τις ευρωπαϊκές λίστες, να πω ότι μετά από δύο χρόνια συζητήσεων με το Συμβούλιο για τον εκλογικό νόμο μας κατέστησαν σαφές ότι από νομικής πλευράς κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά σε αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης με εξέπληξε που ε, κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιήσουμε και τις 73 έδρες. Η ε, μερική ανακατανομή ε, μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα, συρρήκνωση του Κοινοβουλίου για παράδειγμα. Εμείς συζητήσαμε με πολλούς εμπειρογνώμονες και καταλήξαμε σε συγκεκριμένες ελάχιστες ε, σε ελάχιστα μοντέλα τα οποία όλα προβλέπουν μείωση των εδρών για τις μεσαίου μεγέθους χώρες και αύξηση των βουλευτών, των βουλευτών για τις μικρές και τις μεγάλες. Τώρα αυτό, αν πολιτικά γίνεται ή όχι, είναι άλλο θέμα. Ίσως θα μπορούσε να διευκολυνθεί από μια ε, ανακατανομή, μερική ανακατανομή τουλάχιστον των εδρών του Ηνωμένου Τώρα, θα τα εξετάσουμε όλα αυτά και θα συντάξουμε την πρώτη εκδοχή, την πρώτη εκδοχή της έκθεσης μας. Η κυρίαρχη άποψη είναι η χρήση των 73 εδρών πάντως. Και αυτό θα πρέπει να το περάσουμε ως μήνυμα πριν τις εκλογές. Δεν χρειάζεται να συνοψίσω. Θα δείτε την πρώτη προσπάθεια του, για το, ε, που θα κάνουμε για το κείμενο και θα τη σχολιάσετε. Περνάμε στους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers. Έχουμε μία έκθεση Έχουμε τον εισηγητή μαζί μας. Ε, οι Γιούρι και οι Εκον, η συζητούν το θέμα αυτό. Περιμένω δύο λεπτάκια μέχρι να ξαναπάρετε τη θέση σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι θέλετε να φύγετε, σε περισσότερους σε συμβούλους και βοηθούς απευθύνομαι, γιατί από εκεί προέρχεται ε, ο θόρυβος. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να φύγετε ησύχως και να καλέσω τον Φάβιο Καστάλτο που είναι ε, ο εισηγητής για την γνωμοδότηση από πλευρά τη ΑΦΚΟ όπου ξεκινά σιγά σιγά η δουλειά στην Τζούρι και στην ΕΚΟΝ για τα θεμητά μέτρα για την προστασία των πληροφοριδιωτών που ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. Εμεί έχουμε προχωρήσει περισσότερο την εργασία μας από ότι οι αρμόδιε επί τη ουσία επιτροπές. Παρακαλώ συνάδελφοι, ε, εγώ εντάξει να μιλάω με το θόρυβο, αλλά θέλω να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Φάμπιο, αν θες να ξεκινήσεις, θα πρέπει να ξεκινήσεις ε, φωνάζοντας. Ή απλώς θα περιμένουμε δύο λεπτά ακόμα. Those who are already on uh, standing, they don't hear what we are saying. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που στέκονται δεν μας ακούν. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πάλι. Όπως γνωρίζετε σήμερα έχουμε να συζητήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Είναι μια έκθεση της Τζούρι που όμως δεν έχει ε, ακόμα γραφτεί το σχέδιο, πράγμα που βέβαια δεν μας διευκολύνει. Περιμένουμε επίσης ε, να το δούμε για να μπορέσουμε να εκφράσουμε άποψη πιο εμπεριστατωμένη. Ε, έχει δύο εισηγητές, έναν από, το, από τους φιλελεύθερους και έναν από τους σοσιαλιστές. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το θέμα σε αυτήν την χρονική στιγμή και πόσο μου είναι προσφύλες σε μένα προσωπικά αλλά και στο κίνημα των πέντε αστέρων που εκπροσωπώ. Όσον αφορά το κόστος της διαφθοράς στην Ευρώπη, μιλάμε για 218 και 282 δις ετησίως που χάνονται λόγω διαφθοράς. Από αυτά που χάνονται ε, λόγω διαφθοράς, είπαμε. Σε μια περίοδο πολύ έντονης οικονομικής κρίσης, αυτό φυσικά θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ώστε να υπάρξει μια ε, ισχυρή παρέμβαση για την, από πλευρά της Ένωσης για το θέμα των πληροφοριοδοτών, πράγμα που θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Γι' αυτό είμαστε δεσμευμένοι και σε εθνικό επίπεδο, όπου καταθέσαμε την πρώτη πραγματική ε, τέτοια, είδο πρόταση. Επίσης, μέχρι στιγμής είχαμε τομεακή ε, προσέγγιση. Έχουμε εισάγει τέτοιου είδους μέτρα προστασίας ε, των καταγγελτών για συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή τις έμεσες εξουσίες. Όμως, επανειλημμένα το Κοινοβουλίο μας έχει ζητήσει παρέμβαση με πιο γενική προσέγγιση Αναφέρομαι στην έκθεση της Επιτροπής ΚΡΙΜ του 2013 για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος. Αναφέρομαι επίσης στην έκθεση πρωτοβουλία της έκθεσης De Jong της Επιτροπής Κόντ ελέγχου προπολογισμού για το ρόλο των και οικονομικών συμφερόντων στην Ένωση που υιοθετήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 όπου καλείται η Επιτροπή να υποβάλει άμεσα νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο είναι αποτελεσματικό και καθολικό για την προστασία των καταγγελτών και ε, ε, για την πρόληψη των ε, ζημιών εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, πρότεινε να υπάρξει ένας ειδικός θεσμός προστασίας που να τονίζει και να ενημερώνει σε σχέση με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Συνέβαλε και η δική μα Επιτροπή ΔΕ με την εξαίρετη γνωμοδότηση του κυρίου του συναδέλφου Μέσερ Σμιτ. Από την 1η Ιανουαρίου του 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη τη οφείλουν να εισάγουν μέτρα προστασία των πληροφοριδιωτών. Αυτό το έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δηλαδή και το, και το ε, ελεκτικό συνέδριο, ούτε καν δηλαδή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν ε, κάνει το καθήκον τους και η ε, έκθεση Γκίγκολτ για τη διαφάνεια περιλαμβάνει 8 παραγράφους και θυμίζει ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στην ελληνική ομάδα, στην ομάδα Γκρέκο που λειτουργεί στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Τώρα εμείς συζητάμε και την νομική βάση για να υπάρχει μια τέτοια καθολική προσέγγιση για τους πληροφοριοδότες, γιατί ακριβώ αυτό το πρόβλημα ότι είναι αρκετά και κατακαιρματισμένη προσέγγιση και η συζήτηση έχει επικεντρωθεί σε διάφορες επιλογές. Το πρώτο να συνδεθεί με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δηλαδή δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Ε, το δεύτερο είναι να ε, προσεγγίσουμε τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της ε, ενιαίας αγοράς, ε, να ενταχθεί εκεί ένα τέτοιο όργανο, αλλά εκεί αποκλείονται πλαίσια τα οποία βγαίνουν από το πλαίσιο της αγοράς, η εναρμόνιση της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να μπορούν όλοι με τρόπο ελεύθερο να εργάζονται, αλλά αυτό θα, θα κάλυπτε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα και θα ήταν ίσω λίγο πιο ρηψοκίνδυνη η νομική βάση σε σχέση με τα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Και ενδεχομένω υπάρχει και το άρθρο 82, παράγραφος 1, ε, γράμμα D, που μιλάει για δικαστική ποινική συνεργασία ε, σε θέματα ποινικού δικαίου δηλαδή και επιτρέπει και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και δικαστικών αρχών αυτών για την, ε, τα ποινικά δικήματα και για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων από μια μελέτη που έγινε από την Transparency International το 2013 έχουν τεθεί κάποια πρότυπα για την προστασία των πληροφοριοδοτών που αφορούν την καθορισμό κατηγοριών, απαιτεί συγκεκριμένε και σύνολα και ασφαλή κανάλια για την ε, κάζοτε καταγγελία, έπειτα αποδείξεις ε, και έλεγχος του κατά πόσο λαμβάνονται μέτρα ή όχι κατά των ε, πληροφοριοδοτών λόγω του ότι έδωσαν αυτές τις πληροφορίες ε, κάποια πράγματα είναι, ε, καθώς πρόκειται για μια δύσκολη ανθρώπινη επιλογή θα πρέπει να υπάρχει και ψυχολογική προστασία, η στήριξη για την δεχόμενη ανέβρεση νέας θέσης απασχόλησης κτλ. Από αυτή τη μελέτη της ε, Transparency International του 2013 φαίνεται να επικρατεί πολύ διαφορετική κατάσταση ένα κράτος. Αν συγκρίνουμε τα 28 και μελλοντικά 27 κρατή-μέλη, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή στη Ρουμανία, στη Λογανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λουξεμβούργο. Μεσαίου τύπου προστασία στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Δανία, την Εστονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετωνία, τη Μάλτα, την Πολωνία και την Σουηδία και σχεδόν ε, απουσία προστασία στη Βουλγαρία, Φιλανδία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να ορίσουμε μια καθολική προσέγγιση, κοινή προσέγγιση για να προστατεύσουμε τις αξίες της Ένωσης, αυτές που ορίζονται από το άρθρο 2. Διαπιστώνουμε ότι, ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή ε, ε, ίσως βάση, αλλά πρέπει να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες ε, ε, Φάβιο, παρακαλώ να μιλήσεις λίγο πιο αργά, γιατί από ό,τι φαίνεται ε, δυσκολεύονται οι ε, διερμηνείς. Ναι, δεν πειράζει, τέλειωσα. Για να βρούμε μια κατάλληλη νομική βάση, λοιπόν, που να συμφωνεί με τους στόχους που εμείς επιδιώκουμε, που θέλουμε να είναι όχι γίνεται πιο ευρύ και αποτελεσματική. Ελπίζω ότι το σχέδιο της ε, Τζούρι θα υποβληθεί γρήγορα για να μπορέσουμε να μπούμε και στις τεχνικές λεπτομέρειες του ζητήματος με αυτή την πρώτη ανταλλαγή. Εγώ θέλησα μόνο να σταθώ στη γενική εικόνα, στη γενικότερη εικόνα και ε, περιμένω με χαρά τις παρατηρήσεις των σκιωδών και των συναδέλφων που θέλουν να κάνουν προτάσεις ε, και κρίσεις, αναμένοντας, όπως είπα, την δυνατότητα να περάσουμε σε πιο τεχνική τα θέματα. Και ε, πρώτη δηλαδή απόψεων θα έλεγα ότι είναι καλό να ορίσουμε στις 12 Ιουλίου, αν συμφωνείτε όλοι. Ευχαριστώ και πάλι. Thank you. Mm-hmm. Thank Ευχαριστώ πολύ. Κύριε για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να παρέμβω στο όνομα του ΕΛΚΑ για αυτό το σημαντικό θέμα. Καθώς είμαι και μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, γνωρίζω ποιες είναι οι δυσκολίες ε, ε, ολοκλήρωσης ε, του διατακτικού για την εφαρμογή αυτών των εργασιών, την υλοποίηση μάλλον των εργασιών. Καθώς και θα πρέπει ακόμα να καθοριστούν να αποφασιστούν οι εργασίες συνεννόησης για να ξεκινήσουμε την εργασία στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που στόχο έχουν διάφορα θέματα και βέβαια αυτός θα είναι και ο στόχος αυτής της έκθεσης εδώ, όπως και στις άλλες επιτροπές. Όπως είπα, στόχος είναι το βασικό, βασικό ε, ουσιαστικό θέμα της νομικής βάσης επί της οποίας θα βασιστεί ένα κείμενο, σχέδιο μάλλον νομοθετικού κειμένου. Η ομάδα μας, το ΕΛΚΑ, θα είναι πλήρες μέλος, επικοδομητικό, θα συμμετέχει πλήρως στη συζήτηση και στον προβληματισμό, ώστε να μπορέσουμε όντως να προχωρήσουμε σε ένα με πνεύμα βολοταριστικό, σοβαρό, ρεαλιστικό και στις ευθύνε ώστε να φτιάξουμε μια γενική προσέγγιση που θα προχωρεί σε όσο γίνεται πιο εναρμονισμένη προστασία των πληροφοριοδοτών. Είτε πρόκειται για τις εργασίες και τα πορίσματα της Επιτροπής LuxLeaks, της οποίας προέδρευε ο Λέν Λαμασούρ, όσο και σχετικά με την εργασία της Επιτροπής σε Panama Papers, της οποίας προεδρεύει ο Μπέρναντ Λάγκεν. έχουμε δει και αναγνωρίσει τη σημασία του ρόλου των πληροφοριοδοτών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι αποκαλύψεις από το δύο σκανδάλων, το LuxLeaks και το Panama Papers, δεν θα είχαν συμβεί χωρίς να έχουν υπάρξει πληροφοριοδότες. Και μάλιστα ορισμένοι είναι στο στόχαστρο και είναι θύματα, έχουν πολλά προβλήματα και ορισμένοι μάλιστα διώκονται και δικαστικά και έχουν και καταδικαστεί. Εμείς αυτό το καταγγέλουμε και το καταδικάζουμε. Ε, και μάλιστα είχα την ευκαιρία να το κάνω, εργαζόμενοι για την οδηγία που αφορά την προστασία των όσων λέμε ε, ότι είναι επιχειρηματικά μυστικά. Έχουμε γράψει σε ένα ε, νομοθετικό κείμενο και μία διάταξη προστασίας των πληροφοριοδοτών μέσω των εξαιρέσεων. εφόσον αυτοί οι πληροφοριδότες έχουν αναγκαστεί να αποκαλύψουν ένα επιχειρηματικό μυστικό στη διάρκεια της αποκάλυψης ε, στοιχείων που θίγουν το ευρωπαϊκό συμφέρον. Στόχος μας λοιπόν θα είναι να είναι ρεαλιστικό και λογικό αυτό το πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ε, διαφάνεια προς διαφάνειας. Θέλουμε να φτιάξουμε λειτουργικές διατάξεις που να μπορούν να μεταγραφούν εύκολα εάν εγκριθούν από εμά με ισορροπημένο τρόπο στις νομοθεσίες των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ε, Ραμόν Χαουρέγγι τους τους Ο Ραμόν Χαουρέγγι για τους ε, Και εγώ θέλω να εκφράσω την προθυμία μας να συνεργαστούμε με τον κύριο Καστάλτο ως πολιτική ομάδα. Όλοι συμφωνούμε πως το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα είναι σημαντικό. Και εγώ ε, ήμουν μέλος των Επιτροπών τάξη 1, τάξη 2, Panama Papers και έχω έρθει σε επαφή με τους ε, καταγγέλλοντες τις λειτουργίες ε, και οι επαφές αυτές ήταν πραγματικά πολύ φορτισμένες συναισθηματικά. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε εδώ ότι χρειαζόμαστε κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους των οποίων συνεισφορά στο δημόσιο συμφέρον τους οδηγεί, μερικούς τουλάχιστον από αυτούς, να θέσουν σε κίνδυνο την επαγγελματική τους καριέρα, αλλά και τη ζωή τους καμιά φορά. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που συμφωνούμε επί του στόχου, ε, αντιμετωπίζουμε σημαντικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Προστασίας το πρώτο που θα πρέπει να αποφύγουμε για παράδειγμα είναι ε, αυτές οι συμπεριφορές να χαρακτηρίζονται ως αδικήματα και ε, ως ποινικά αδικήματα πολλές φορές χαρακτηρίζονται. Και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ε, ε συστήματα της ε, ενομιστάξης ε, των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος ε, έχει τις δικές του αρμοδιότητες και δεν δέχονται τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους υπαγορεύσει ε, ποια μορφή θα πρέπει να πάρει ο ποινικό του κώδικας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η ε, οδηγία την οποία ζητούμε εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που ήρθε στην επιφάνεια το σκάνδαλο LuxLeaks, το Κοινοβούλιο τα να τους ε, προστατεύσει, αλλά ο Αντουάν Τελτούρ καταδικάστηκε τελικά, το οποίο σημαίνει ότι η προστασία είναι λυπής. Και η οδηγία, λέω, την οποία ζητούμε εδώ και καιρό, θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιες παρεμβάσεις στους δεοντολογικούς κώδικες ε, ε, ή στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών. Ε, Λέω πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσει και μηχανισμού που να είναι αποτελεσματικοί. Η Κομισιόν ξεκίνησε μια διαβούλευση που ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου. Είναι σημαντικό αφενός η Κομισιόν να μας ενημερώσει για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης που ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου. Παράλληλα όμως η κυρία Βερστάγκερ δημιούργησε ε, ένα σύστημα το οποίο μου φαίνεται πολύ αποτελεσματικό που είναι ε, το ανώνυμο ε, σύστημα καταγγελιών. Ένας υπάλληλος μιας ε, τράπεζας ή μιας ενός κεφαλαίου ή ενός σηματοπιστωτικού ιδρύματος κλπ. μπορεί να αναγγείλει πράγματα τα οποία ε, είναι, ε, βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον με ανώνυμο τρόπο χωρίς δηλαδή να διακινδυνεύσει τίποτα. Ε, αυτό διευκολύνει πολύ την κατάσταση. Ίσως είναι ένα καλό σύστημα. Και από τις 22 Μαρτίου η κυρία Φερστάγκερ είπε όποιος ε, θεωρεί ε, ότι ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές ε, δεν είναι κατάλληλες μπορεί να τις καταγγείλει με πλήρη μυστικότητα και χωρίς αποκάλυψη ταυτότητάς του. Ίσως να είναι καλό αυτό και ίσως ένα τέτοιο μηχανισμό χρειαζόμαστε. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει ενδεχομένως να ε, προστατεύουν την εμπιστευτικότητα τέτοιων καταγγελιών. Αλλιώς ε, κινδυνεύουν ε, από τα συστήματα, τα ένωμη τάξεις των κρατών μελών να καταδικαστούν ε, για τις καταγγελίες αυτές. Αυτά, επαναλαμβάνω, είμαστε αναφαντών υπέρ τη συνεργασία με τον κύριο Καστάλτο ε, και κατά τα άλλα θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μάιτε για το Άλτε. Θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο κύριος Χάουρεγγι. Και εμείς ε, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τον κύριο Καστάλτο. Είμαστε σίγουροι θα η εργασία του θα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω αν μάθατε ότι το βραβείο Πούλιτζερ τον, το κέρδισε το Διεθνές Κονσόρτσιο που ε, ε, έφερε στο φως της δημοσιότητας ε, το σκάνδαλο των Panama Papers. Εμείς εν μεταξύ έχουμε μια ειδική επιτροπή διαρεύνησης και ευτυχώς για τον κύριο Ντό δεν ήξερε ποιος ήταν. Ο, το άτομο το οποίο δημιούργησε αυτή την αναστάτωση σε διάφορα σημεία του πλανήτη που προκάλεσε έρευνες στη δική μας επιτροπή κλπ. Ε, ε, δεν θα είχε, δεν θα ήταν τόσο προστατευμένος αν είχε γίνει γνωστή ταυτότητά του. Εγώ γνώρισα προσωπικά ένα άτομο το οποίο στην Ισπανία κατήγγειλε συγκεκριμένες δυσλειτουργίες και ε, όχι μόνο έχασε τη δουλειά του, Ε, και ήταν και πολύ ισχυρή ε, στην περιοχή στην οποία ζούσε, όμως μπήκε σε μια μαύρη λίστα, σε ένα μαύρο κατάλογο ε, και σχεδόν καταστράφηκε η ζωή της. η πολλά εγκλήματα τα οποία σχετίζονται με διαφθόρα, με τις λειτουργίες κλπ. κλπ είναι και διασυνοριακά. Ακόμα και η προσωπική αντίληψη του καθενός για το τι είναι αδίκημα και έγκλημα διαφέρει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ναι, όλοι μαζί να κάνουμε αυτή τη δουλειά στη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Μαξ Άντερσον. Θέλετε το λόγο? Όχι. Γιατί είναι το όνομά σα στον κατάλογο μιλτών. Αλλά δεν θέλετε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά παρόλα αυτά παραμένετε σκιώδη. Ωραία. Κανεί άλλο δεν θέλει το λόγο. Πρώτη φορά στην Επιτροπή μας εκφράζεται αυτή η διάθεση επικοδομητικής συνεργασίας. Δεν ξέρω, Φάμπιο, τι τους έχεις κάνει και τους μάγεψες. Παρ' όλα αυτά, σε συγχαίρω. Στην Γιούρη εκκρεμεί ακόμα ο διορισμός ε, των ε, συνεισηγητών, γι' αυτό και έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο. Επόμενη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει τον Ιούλιο στις 12 του μηνός και μετά στο τέλος του Αυγούστου θα δούμε τις τροπολογίες και τελική ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Αλλά θα έχουμε μια ευελιξία βάσει και ε, του πώς θα προχωρήσει το, η δουλειά αυτή στις Επιτροπές Γιούρη και Έκον. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο ξανά σε σένα για να κάνεις τελικές σου παρατηρήσεις. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Ε, Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τους προλαλήσαντες για, τη, για τα λόγια τους, για τη συνεργασία την οποία είναι πρόθυμοι να προσφέρουν. Ευχαριστώ επίσης και τους γαλλόφωνους συναδέλφους Ε, αυτά που είπατε για το LuxLeaks και το σκάνδαλο των Panama Papers ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Χρειάζεται να αντιδράσουμε πολιτικά καταρχήν. Γιατί οι πολίτε έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό ακριβώς διότι δεν βλέπουν ε, και άμεσες απαντήσεις στα προβλήματά τους. Ελπίζω σύντομα να έχετε το... Ε, ελπίζω σύντομα να έχουμε στα χέρια μας την πρώτη έκθεση της Γιούρη, το προσχέδιο, αλλά νομίζω ότι ε, σε ό,τι αφορά τη νομική βάση θα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες μας, την, ε, το, το, το περιθώριο που μας δίνει ο νόμος και την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τα σκάνδαλα είναι αποδεδειγμένα. Η αλήθεια έχει λάμψει. Οπότε από ηθικής πιο πολύ πλευράς και όχι μόνο πολιτικής δεν είναι δυνατόν οι υπεύθυνοι, να μην τιμωρούν, να, ε, δεν είναι δυνατόν, συγγνώμη, οι καταγγέλλοντες να τιμωρούνται στην εθνική δικαιοσύνη της α της Νομίζω ότι οι συζητήσεις θα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες. Ε, εγώ δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ καλά με όλους και με όλες σας. Ελπίζω θα καταλήξουν σε καλές συμβαστικές λύσεις που ελπίζω ότι θα προβάλλουν μια ισχυρή φωνή από πλευρά του Κοινοβουλίου και μια πραγματική απόδειξη δράσης και όχι μόνο δημιουργίας επιτροπών, διερεύνης κλπ. Νομίζω ότι έτσι θα δώσουμε και ένα δείγμα γραφής ε, ως Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δηλαδή απαντούμε στις ανησυχίες του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ήθελε να τοποθετηθεί. Βεβαίω έχετε το λόγο. Συστηθείτε μα καλώς παρακαλώ. Ναι. Αλεξάνδρα Χέα. Εργάζομαι στην ε, ε, στο τμήμα C2 της DigiJust ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να πω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει στεναρά τον στόχο της προστασίας των πληροφοριοδοτών και έχει αναλάβει βήματα προκειμένου να προστατεύει ε, τους πληροφοριοδότες στην κλαδική ενωσιακή νομοθεσία και στην ανακοίνωση της 5ης Ιουλίου 2016 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ε, θα εξετάσει ε, την δυνατότητα ανάληψης κλαδικής οριζόντιας δράσης για την προστασία των πληροφοριοδιωτών, σεβόμενη βεβαίως την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα εργασιών για το 2017, η Επιτροπή ε, εκτελεί μελέτη αντικτύπου η οποία ξεκίνησε και ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου μια δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση η οποία θα είναι ανοιχτή έως τις 29 Μαΐου. Και η μελέτη και η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν την Επιτροπή προκειμένου να εξελογήσει την, ε, τον βαθμό που χρειάζεται κλαδική οριζόντια νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η μελέτη που εκπονεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη, συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών. Τα αποτελέσματα της μελέτης και της διαβούλευσης θα δημοσιευθούν τον ε, Ιούλιο του 2017 τα οποία και θα μας επιτρέψουν να λάβουμε μια ενημερωμένη απόφαση σχετικά με την πολιτική ή την νομοθετική πρωτοβουλία που θα αναλυφθεί σε ενωσιακό επίπεδο, σεβόμενη, βεβαίως όπως είπα πάντοτε την αρχή της επικορικότητας και θα εξετάσουμε ποια ε, μέτρα θα μπορούσαν να κριθούν κατάλληλα. Όπως είπα, μπορεί να πρόκειται είτε για ε, βήματα πολιτικής, είτε για οριζόντια, είτε για κλαδική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Να κλείσουμε αυτό το θέμα. Να ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 2 και 3 Μαΐου. Ε, θα είναι στις, ε, την, ε, την, ε, την Δευτέρα Μαΐου θα είναι ε, μικρή η απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Τίμερ, Τίμερμαντς και θα έχουμε και την διακοινοβουλευτική συνάντηση. Θα έχουμε δηλαδή εκπροσώπους Εθνικών Κοινοβουλίων εδώ σχετικά με την εφαρμογή των ε, με την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης που αφορούν τις ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών, οπότε όποιοι δεν έχουν δουλειά, παρακαλώ να αποχωρήσουν την αίθουσα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.